αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να σας καλωσορίσω σε αυτή τη κοινή συνάντηση της Δεκάμπ με την ομάδα παρακολούθησης της ΣΥΝΤΡΑ για την Κεντρική Αμερική. Θα καλωσορίσω επίσης τον συμπρόεδρο αυτής της συνάντησης, τον κύριο Μπόγκε, και τους αντιπροέδρους της αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με την Κεντρική Αμερική. Θα ήθελα να καλωσορίσω θερμά τους επισκέπτες μας, τον κύριο Αλεξάνδρ Μόρα, Υπουργό Εξωτερικού Εμπορίου της Κωνσταντίνα, την κυρία Μαρτσέλα Τσαβαρία, Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εξωτερικού Εμπορίου της Κωνσταντίνα. Θα ήθελα επίσης να καλωσορίσω όλους τους εκπροσώπους των διπλωματικών αποστολών και ιδίως στην αυτοεξοχότητα τον κύριο Αλφάρο, πρέσβη της Κωνσταντίνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τον κύριο Αλεχάνδρο Πατίνο, επικεφαλή του εμπορίου του Γραφείου Διασύνθεση του Υπουργείου Εξωτερικού Εμπορίου τη Κωνσταντίνα για τι υποθέσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΟΣΑ, να καλωσορίσω επίσης τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, τον κύριο Φερνάντε Πόνς, ο οποίος θα έρθει σε λίγο όπως μας έχει ειδοποιήσει. Να σας πω ότι η διερμηνία θα παρέχεται στις εξής γλώσσες που είναι τα αγγλικά, τα ισπανικά, τα ελληνικά και τα ιταλικά. Σας έχει διανεμηθεί η ημερήσια διάταξη στα αγγλικά, στα ελληνικά και στα ισπανικά και αν δεν υπάρχει κάποια αντίρρηση μέχρι το τέλος της συνεδρίασης θα επικυρωθεί όπως έχει. Και θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Μπόγκε που μας πει δύο λόγια. Thank you very much, uh, Mr. President. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι. Είναι μεγάλη μας χαρά που σήμερα θα έχουμε αυτή την ευκαιρία να από απόψεων μαζί σας. Ακριβώς, όπως έγινε και με την ομάδα παρακολούθησης για το εξωτερικό εμπόριο. Πριν από κάποιους μήνες και έτσι θα εξετάσουμε τις ε, προτεραιότητες της Προεδρίας. Έχουμε τρεις-τέσσερις σημαντικές ερωτήσεις που μας ενδιαφέρουν και θέλουμε να ακούσουμε την άποψή σας όσον αφορά τις πρόσφατες εξελίξεις στα εμπορικά θέματα Θέλω να δούμε τι γίνεται με την κατάσταση στην ΣΥΑΚΑ και επίσης να μας πείτε με δύο λόγια πώς προχωρούν οι διαπραγματεύσεις, να μας πείτε τι προβλήματα αντιμετωπίζετε, γιατί όπως και στην Ευρώπη και εκεί υπάρχουν πολλές διαφορετικές χώρες με διαφορετική διάρθρωση, δομή και άρα αυτό έχει σαν αποτέλεσμα διαφορετικές συνέπειες για την πολιτική στα εμπορικά θέματα. Επίσης έχουμε και την τελωνιακή συμφωνία και αυτό μας ενδιαφέρει να ακούσουμε τη δική σας γνώμη και ποιες θεωρείτε ότι είναι οι κορυφαίες προτεραιότητες της Προεδρίας. Επίσης, η επόμενη Προεδρία θα ανερθεί από τον Πανάμα. Οπότε να μας πείτε ακριβώς πώς θα συναρθρωθείτε, αν έχετε κάποια, κάποιο κοινό θεματολόγιο, ε, αν μπορείτε να μας ενημερώσετε. Κάτι άλλο τώρα. Με μεγάλο ενδιαφέρον παρακολουθήσαμε τις προσπάθειες που καταβάλατε για να γίνετε μέλος του ΟΣΑ. διαβάσαμε τα σχετικά έγγραφα με προσοχή. ξεκίνησε αυτή η διαδρομή το 2015. Ήδη έχουν γίνει 22 αξιολογήσεις για την προσχώρησή σας, αλλά εδώ ε, είναι η πρώτη ευκαιρία που το συζητούμε. Άρα βλέπουμε ότι σε αυτό το μέτωπο προχωράτε πιο γρήγορα από ότι σε άλλους τομείς. Τώρα για να δούμε ε, τι θα γίνει τώρα που ανέστηλε τη συμμετοχή στην TTP ο πρόεδρος Τραμπ για να δούμε τι γίνεται όσον αφορά την ε, διακοπή και αναστολή ισχύω των εμπορικών συμφωνιών και να δούμε ποιες είναι συνέπειες για τις δικές σας εμπορικές δραστηριότητες για την λεγόμενη ε, συμμαχία του ειρηνικού και ε, να δούμε ποιες είναι οι συνέπειες για τη συμφωνία σύνδεσης για τον σχετικό πυλώνα και την εφαρμογή αυτού. Βεβαίως και εδώ θα πρέπει να έχουμε κριτική θεώρηση του τι έχουν κάνει τα κράτη-μέλη. Αλλά αυτό δεν είναι δικό σας θέμα. Ε, φταίτε εσείς. Πολλές φορές έχουμε ε, πολύ αργή κύρωση των συμφωνιών σύνδεση από πλευρά κάποιων εθνικών κοινοβουλίων και θυμάμαι ότι πριν από κάποιους μήνες είχαμε εδώ τον πρέσβη της ε, Γουατεμάλα και μιλούσαμε για τη σχετική ομάδα παρακολούθηση και μας έλεγε ότι και αυτός αντιμετώπιζε ένα τέτοιο πρόβλημα. Πάντως δεσμευόμαστε να τα πούμε όλα αυτά στους επικεφαλείς του Κοινοβουλίου και έτσι να επιταχυνθούν οι συνομιλίες με τα κρατημέλια για να δούμε τι θα γίνει στο μέλλον ούτως ώστε να μην χαθεί η αξιοπιστία. Χρειάζεται να υπάρξει αυτή η διαδικασία κύρωση. Να μην έχουμε αυτή τη διαδρομή των τριών ετών. Δεν είναι σωστή συμπεριφορά. Καλώς ορίσατε επομένω και ευχαρίστω να σας ακούσουν. Γεια σας. Καλώς απόγευμα. Αγαπητή κυρία Σακοράφα, πρόεδρε της ε, αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με τις χώρες της Κεντρικής Αμερικής, ε, κύριε Μπέργκε, από την ομάδα παρακολούθησης της Επιτροπής ΣΥΝΤΑ για τη Συμφωνία Σύνδεσης Κεντρικής Αμερικής ευρωπαϊκή Ένωσης. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, αγαπητοί πρέσβεις φιλικών χωρών, κυρίες και κύριοι υπάλληλοι των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διπλωμάτες, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή Ίντα και την ΔΙΚΑΜ, την Αντιπροσωπεία της σχέσης με τις χώρες Κεντρικής Αμερικής, που μου επιτρέπουν να είμαι εδώ σήμερα και να σας ενημερώσω για τις εργασίες της Κώστα Ρίκα, ε, όπως αυτές εξελίσσονται τα τελευταία χρόνια. Και να σας ενημερώσω επίσης για το τι θα κάνουμε τους επόμενους μήνες. Βρίσκομαι εδώ σήμερα όχι μόνο ως ε, Υπουργός Εξωτερικού Εμπορίου της Κωνσταντίνα, υπεύθυνο για τις σχέσεις, ε, εμπορικές σχέσεις Κωνσταντίνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε μόνο ως συντονιστής της διαδικασίας της ένταξης Κωνσταντίνα στον ΩΣΑ, αλλά και ως πρόεδρος, ε, προσωρινός πρόεδρος του Συστήματος Οικονομικής Ολοκλήρωσης τη Κεντρικής Αμερικής, της ΣΥΕΚΑ. Θα ήθελα λοιπόν να σας μιλήσω για τρία ζητήματα. Πρώτον, το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η εφαρμογή του εμπορικού πυλώνα της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κεντρικής Αμερικής. Δεύτερον, για το πρόγραμμα ε, της προσωρινής, εργασία προσωρινής προεδρίας του συστήματος ολοκλήρωσης ε, της Κεντρικής Αμερικής, η Κωνσταντίνα προεδρεύει το πρώτο εξάμεινο και ο παναμά το δεύτερο εξάμεινο του 2007. Τρίτον, για το στάδιο και την πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε ό,τι αφορά την ένταξη της Κωνσταντίνα στον ΟΣΑ και ορισμένα, θα σας μιλήσω και για ορισμένα από τα στοιχεία για τα οποία έκανε ερωτήσει ο κύριος Μπέγκε. Σε ό,τι αφορά τη συμφωνία σύνδεσης ε, μεταξύ Κεντρικής Αμερικής και Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί ένα στοιχείο κλειδί της ε, διεύρυνσης και της εμβάθυνσης της εμπορικής πλατφόρμας της ε, χώρας μας και αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία ανάπτυξης για την Κεντρική Αμερική. Η εφαρμογή της Συμφωνίας Πλαίσιο αποτελεί ε, το ξεκίνημα μιας πιο πλατιάς και πιο βαθιάς σχέσης ε, ε, μεταξύ των δύο περιφερειών. το, η ροή των, η εμπορική ροή της Κωνσταντίνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση έφτασε στο 82,6% των συνολικών εισαγών και το 84,9% των συνολικών εξαγών. Όχι με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με όλες τις άλλες τρίτες περιοχές του πλανήτη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι παλιός ε, φίλος και σύμμαχος ε, και το εμπόριο με την Ευρωπαϊκή Ένωση αντιπροσωπεύει το 12,9% του συνολικού εμπορίου της Κωνσταντίνα για το 2015. Για φέτος το 18,5% των εξαγωγών μας ε, πήγαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το 9,4% των εισαγωγών μας προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την τελευταία δεκαετία οι εμπορικές μας σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ε, θετικό ισοζύγιο ε, και αναπτύσσονται κατά μέσο όρο με 2,5, ε, κατά 2,5% κατ' Ε, μια αλλαγή στην δομή των εξαγών της Κωνσταντίνα, καθώς επίσης και κάποιες κλιματικές αναταραχές που εμφανίστηκαν έχουν επηρεάσει τις στατιστικές των τελευταίων ετών, κάτι που δεν μας επιτρέπει να αξιολογήσουμε το αποτέλεσμα της Συμφωνίας Σύνδεσης από όταν τέθησε ισχύ. Παρ' όλα αυτά, αν εξαιρέσουμε αυτά τα ε, συγκυριακά στοιχεία, οι εξαγωγές ε, προϊόντων από την Κωνσταντίνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν τάση αύξησης. Ε, κυρίως σε τομείς που ενδυναμώθηκαν πολύ, όπως για παράδειγμα οι ιατρικές, ο ιατρικός εξοπλισμός, εξοπλισμός ακριβίας, των οποίων οι εξαγωγές ε, προς την Ευρωπαϊκή Ένωση φτάνουν στο 24% του συνόλου των εξαγωγών μας. Είναι σημαντικό, σημαντική αύξηση. Η διμερής ε, σχέση μας επίσης έχει σημαντικό δυναμικό για το μέλλον και σημαντικές ευκαιρίες στο επίπεδο των επενδύσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, κάνει τα τελευταία δέκα χρόνια το 18% των άμεσων ξένων επενδύσεων που δέχεται η Κωνσταντίνα ε, και μάλιστα σε τομείς ε, που διαφοροποιούνται και σε καινούριου κλάδους που έχουν σχέση με την τεχνολογία και την καινοτομία. Στο πλαίσιο της Συμφωνίας Σύνδεσης και τις ιδιαίτερες σχέσεις που διατηρούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση ελπίζουμε ότι θα συνεργαστούμε και στο μέλλον για την ε, πλήρη εφαρμογή της Συμφωνίας Σύνδεσης με στόχο να εξασφαλίσουμε ότι θα εκμεταλλευτούμε πλήρως τις ευκαιρίες που δημιουργούνται. Τώρα, σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα εργασίας της ε, προσωρινής Προεδρίας του Συστήματος Οικονομικής Ολοκλήρωσης της Κεντρικής Αμερικής, την οποία αυτή τη στιγμή έχει αναλάβει στο πρώτο εξάμεινο η Κώστα και στο δεύτερο εξάμεινο Παναμάς. Το Συμβούλιο Υπουργών της ε, ε, ΣΥΕΚΑ το Κομιέκο δηλαδή, υιοθέτησε το πρόγραμμα δράσης για τη διαδικασία της Τελωνικής Ένωσης, ε, ε, του οποίου ηγείται η Κωνσταντίνα το πρώτο εξάμεινο και το Παναμά το δεύτερο εξάμεινο. Με αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλίσουμε την συνέχεια και ελπίζουμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα επιταχύνουμε μια σειρά εργασιών που εκκρεμούν. Μεταξύ των πρωτοβουλειών που θα, πρέπει, που θα σκοπεύουμε να προωθήσουμε είναι να προχωρήσουμε ε, στην ε, συμμόρφωση με τις δεσμεύσεις που αναλάβαμε στο πλαίσιο της Συμφωνίας Σύνδεσης και ε, των δεσμεύσεων που προκύπτουν από το πρωτόκολλο ένταξης του Παναμά στο υποσύστημα οικονομικής ολοκλήρωσης. Θέλουμε να προχωρήσουμε σε όλα τα θέματα οικονομικής ολοκλήρωσης και στην δημιουργία και πλήρη λειτουργία της Τελωνιακής Ένωσης στην Κεντρική Αμερική. Σε θέματα όπως η δεσμολογική πολιτική, η εναρμόνιση των τεχνικών κανόνων και οι τελωνιακές διαδικασίες. Σε θέματα διευκόλυνσης του εμπορίου έχουμε κυρίως τη στρατηγική διευκόλυνσης του εμπορίου με έμφαση στη συντονισμένη διαχείριση των ε, σύνορων και στην ε, ψηφιακή πλατφόρμα εμπορίου της Κεντρικής Αμερικής. Αυτή η πλατφόρμα είναι μια οικονομική πρωτοβουλία, καινοτόμως πρωτοβουλία, με τεράστιες ε, δυνατότητες. Έχει ως στόχο ο εξωτερικό, το τομέα του εξωτερικού εμπορίου στην Κεντρική Αμερική να είναι ο πρώτο πλήρω ψηφιοποιημένο τομέα, όπου οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή να μπορεί να γίνει ψηφιακά χωρί την ε, ε, παρέμβαση του ανθρώπινου παράγοντα. Ελπίζουμε ότι αυτό θα μας επιτρέψει να αντιμετωπίσουμε προβλήματα και περιορισμούς που είχαμε στο παρελθόν σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των συνόρων. Αυτό το ε, ηλεκτρονικό εργαλείο, εκτός του ότι θα αυτοματοποιήσει οι διαδικασίες και θα τις επιταχύνει, στις εισαγωγές και τις εξαγωγές, θα μειώσει και τα κόστη. Και εποφελούμε αυτής της ευκαιρίας για να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Ένωση που στήριξε αυτή την πρωτοβουλία και κατέστησε δυνατή την, το ξε, κατέστησε δυνατή το ξεκίνημα αλλά και την ενίσχυση αυτής της διαδικασίας περιφερειακής ολοκλήρωσης που θα μας οδηγήσει σε υψηλότερους, ε, υψηλότερους δείκτες οικονομικής ανάπτυξης και με περισσότερη απασχόληση. Το πρόγραμμα δράσης επίσης περιλαμβάνει την συμμόρφωση με, τους, με τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο της ε, Συμφωνίας Σύνδεσης και ιδιαίτερα εκείνες τις δεσμεύσεις που έχουν προθεσμία 5 ετών όπως για παράδειγμα η εναρμόνιση της ε, τελωνικής νομοθεσίας και οι, τεχνική, οι τεχνικές κανονιστικές ρυθμίσεις. Τέλος, αυτό το εξάμεινο ε, θα ξεκινήσουμε ε, την εφαρμογή του προγράμματος συνεργασίας ΣΥΕΚΑ και όσα στο πλαίσιο του προγράμματος, του περιφερειακού προγράμματος του ΟΣΑ για τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική με στόχο να ενισχύσουμε την τεχνική δυνατότητα της ΙΑΚΑ και του υποσυστήματος οικονομικής ολοκλήρωσης. Με αυτόν τον τρόπο θα στηρίξουμε την ανάπτυξη και την ολοκλήρωση ε, ε, των οικονομικών δυνατοτήτων μας. Μέσω αυτού του προγράμματος η Κώστα Ρίκα θέλει να προωθήσει μια πρωτοβουλία σε επίπεδο κέντρου Λυπικής Αμερικής σε συνέργεια με την ΟΣΑ και τη ΣΥΕΚΑ και με μια ενδεχόμενη οικονομική στήριξη την οποία ζητούμε και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και που νομίζω έχει γίνει το αίτημά μας θετικά αποδεκτό. Ε, με δύο στόχους. Πρώτον, να ενισχύσουμε την θεσμική ε, ανάπτυξη της ε, οικονομικής ολοκλήρωσης μέσω της ε, ε, τη εγκαθίδρυση ενό τεχνικού και πολιτικού διαλόγου μεταξύ ΟΣΑ και ΣΥΕΚΑ. Δεύτερον, την ενίσχυση του ΟΣΑ στην ΣΥΕΚΑ έτσι ώστε αυτή να αποκτήσει καλύτερε ικανότητε τεχνική ανάλυση και αξιολόγηση ε, των κρατικών πολιτικών τη Κεντρική Αμερική σε θέματα όπω το εμπόριο, οι επενδύσει, η, η περιφερειακή ολοκλήρωση, οι υπηρεσίε, η ανάπτυξη τη παραγωγικότητα, η στατιστική ε, και ε, έρευνα. Τέλος, σε ό,τι αφορά το πόσο έχει προχωρήσει η διαδικασία ένταξης της Κωνσταντίνα στον ΩΣΑ. Ε, με χαρά μπορώ να σας ενημερώσω ότι ο πρόεδρος ε, Σολής έθεσε ως στόχο ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης της Κωνσταντίνα στον ΩΣΑ ε, μέσω των 22 επιτροπών στις οποίες εργάζεται η Κωνσταντίνα παράλληλα έθεσε ως προθεσμία το Μάιο του 2018 η ομάδα υπουργών και ε, αξιωματούχων 33 ε, θεσμικών οργάνων της ε, χώρας μας, την οποία συντονίζει το Υπουργείο Εξωτερικού Εμπορίου, εργάζεται σε τεχνικές πτυχές της διαδικασίας, έτσι ώστε να πετύχουμε αυτό το στόχο. Πρόκειται για μια διαδικασία έντονη και εντατική, που απαιτεί σημαντικές και πολλές μεταρρυθμίσεις και εξυγχρονισμό του κράτους και σε διοικητικό επίπεδο αλλά και σε νομοθετικό επίπεδο. Έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο σε αυτή τη διαδικασία αξιολόγησης. Έχουμε ξεκινήσει 21 από τα 22 κεφάλαια αξιολόγησης, ε, τα οποία έχουμε συμφωνήσει με τον ΩΣΑ. Και όπως είπε και ο κύριος βουλευτής, ε, η Επιτροπή Εμπορίου εξέδωσε θετική γνωμοδότηση πολύ πρόσφατα. Ελπίζουμε ότι τους επόμενους μήνες και άλλες επιτροπές ε, θα συνεχίσουν να δίδουν θετικές νομοδοτήσεις έτσι ώστε να προχωρήσουμε. Ε, όλα αυτά αντικατοπτρίζουν την δέσμευση της κυβέρνησης Κωνσταντίνα να ενταχθεί στον ΩΣΑ και να ακολουθήσει τις καλές πρακτικές, να τηρήσει τα τις ψηλές προδιαγραφές του ΩΣΑ ε, και της Ευρώπης γενικότερα. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε στην εφαρμογή των συστάσεων του ΩΣΑ και ελπίζουμε ότι ο δρόμος τον οποίο θα, τον οποίο ακολουθούμε θα μας οδηγήσει στο στόχο μας. Σε ό,τι αφορά την ένταξη ε, στον ΩΣΑ, ε, αυτή έχει και ένα ακόμα στόχο. Θέλουμε ε, να μας επιτρέψει την ανταλλαγή εμπειριών ανάμεσα στον ΟΣΑ και την Κεντρική Αμερική. Αυτό είναι απολύτως απαραίτητο σε μια περιοχή όπου οι ευκαιρίες βελτίωσης είναι τεράστιες και που η ένταξη της στον υπόλοιπο κόσμο αποτελεί τμήμα της οικονομικής ατζέντας. Τελειώνοντας, και ω συμπέρασμα μπορώ να σα πω τα εξή, Η Κωνσταντίνα ε, ποτέ δεν επέτρεψε το μέγεθο της να περιορίσει τις φιλοδοξίε της. Είμαστε μια χώρα μικρή, αλλά με μεγάλες φιλοδοξίε. Το μέγεθός μας ε, δεν ήταν ποτέ εμπόδιο ώστε να τοποθετηθούμε στον κόσμο ε, σε τομείς όπως το εμπόριο, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ειρήνη, η εκπαίδευση ή το περιβάλλον. Αυτές οι αρχές ε, είναι, αυτές οι αξίες, είναι και αξίες της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και βέβαια και των υπόλοιπων χωρών της Κεντρικής Αμερικής. Η Κώστα Ρίκα ε, στην ιστορία της έχει λάβει σημαντικές πολιτικές αποφάσεις, αποφάσεις συγγνώμη, ε, που έθεσαν τα θεμέλια της ταυτότητάς μας ε, και επηρέασαν σε βάθος της, το μετασχηματισμό της κοινωνίας μας αλλά και της κοινωνίας των υπόλοιπων χρόνων της Κεντρικής Αμερικής. Αυτή η ηγετική μας ε, θέση διατηρείται εδώ και πολύ καιρό προσπαθώντας και ενθαρρύνοντας μια Κεντρική Αμερική πιο δυναμική, πιο δίκαιη και πιο συμμετοχική παρόλο ότι η χώρα μας και η Κεντρική Αμερική έχει, έχουν κάθε μία τις δικές, τους, τις δικές της προκλήσεις, εμείς στην Κωνσταντίνα θέλουμε να συνεχίσουμε τις επιτυχίες μας. Και γι' αυτό λόγο ε, έχουμε πάρει σημαντικές αποφάσεις. Η συμφωνία Σύνδεσης τη Κεντρική Αμερική με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα καλό παράδειγμα. Η Κώστα είναι μια χώρα που έχει εστιάσει την ανάπτυξή της ε, ε, στη λογική της ε, ολοκλήρωσης καθώς επίσης και του σεβασμού της πολυμερούς προσέγγισης. Αυτή η εστίαση είναι πολιτική, κρατική πολιτική, κρατική επιλογή στην Κωνσταντίνα και θα συνεχιστεί. Γνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή έχουν προκύψει ιδιαίτερες συνθήκες στη διεθνή σκηνή. Ξέρουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν λάβει μια σειρά αποφάσεων, τουλάχιστον έχει ανακοινώσει κάποιες αποφάσεις που θα ληφθούν στο μέλλον. Ε, το σεβόμαστε, τι σεβόμαστε αυτές τις αποφάσεις, αλλά είμαστε ξεκάθαροι. Η Κώστα Ρίκα θα συνεχίσει να επιμένει στην σημασία της ολοκλήρωσης, στη σημασία της οικονομικής απελευθέρωσης ως εργαλείο ανάπτυξης και στην σημασία πολυμερών προσεγγίσεων ε, και πολυμερούς διακυβέρνηση σε όλα τα όργανα στα οποία συμμετέχουμε. Θέλουμε να ενισχύσουμε αυτή την προσέγγιση και το ίδιο ελπίζουμε και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε και από τη δική μας πλευρά να συνεισφέρουμε συνεχώς στην ανάπτυξη των δυνατοτήτων ολοκλήρωσης. Και αυτή τη στιγμή είμαστε εδώ για να επαναλάβουμε αυτή την προσήλωση της Κωνσταντίνα στην ε, ε, ολοκλήρωση, στην ανάπτυξη, στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην πρόοδο ε, υπέρ των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του, των Ηνωμένων Εθνών και για να επαναλάβουμε μία ακόμα φορά την προσήλωση να εργαστούμε σε όλη μας την περιοχή της Κεντρικής Αμερικής προκειμένου να προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση και στη σχέση μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμμαχο και φίλο. Ε, η Κεντρική Αμερική είναι μια περιοχή ανοιχτή που προωθεί τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ειρήνη και τις κοινέ μας αξίες. Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω ευχόμενος το καλύτερο και δηλώνοντας ότι είμαι στη διάθεσή σας να συνεργαστούμε στενά. Θα ήθελα να επαναλάβω τις ευχαριστίες μου και ελπίζω ότι θα στηρίξετε όλες και όλοι εσείς την διαδικασία την οποία αυτή τη στιγμή συντονίζουμε και της οποίας ηγούμεθα για την οικονομική ολοκλήρωση της Κεντρικής Αμερικής. Ευχαριστώ. Και εμείς σας ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ για τις τόσο σημαντικές πληροφορίες που μας δώσατε και τώρα θα ήθελα να ρωτήσω τον αναπληρωτή επικεφαλή της μονάδας στην ε, εξωτερικής δράσης για την Κεντρική Αμερική, το Μεξικό και την Καραϊβική, τον κύριο Πόνσε, αν θέλει να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, και πολλές ευχαριστίες προς τον κύριο Υπουργό για την ε, παρουσίαση που έκανε και θα πρέπει Πρώτα-πρώτα να πω ότι συμφωνώ με τη δεσμευσή του, τόσο ώστε οι κοινέ αξίες να προωθηθούν, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η προστασία του περιβάλλοντος, οι στόχοι της βιώσιμης ε, ανάπτυξης, γιατί είναι πολύ σημαντικά, όπως και η καταπολέμηση της περιθωριοποίησης. Οπότε και όλα αυτά ε, μας βρίσκουν συμφώνους και το υποστηρίζουμε. Επίσης, θα πρέπει να πω προ Βορρά και προς όλου τους ε, εταίρου μα, ότι συμφωνούμε με όσα είπε ο κύριο ε, υπουργό για το ότι τώρα έχουμε μια ευκαιρία για να είναι πιο καλή, πιο πλήρης η συνεργασία μας. Οπότε θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με την εφαρμογή του εμπορικού πυλώνα. Αυτό είναι σημαντικό και για μας και για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Παρ' όλα αυτά θεωρούμε ότι θα βοηθήσει η Κωνσταντίνα με την Προεδρία της, αλλά και με το ότι θα τηρήσει τις δεσμεύσεις της, όπως είπε ο κύριος υπουργό. Και έτσι θα επικαιροποιηθούν αυτές οι συμφωνίες όσον αφορά την ιδιότητα του μέλους και θα βοηθήσουμε ούτως ώστε να έχουμε συνεργασία όλο και πιο στενή στα εμπορικά θέματα. Τώρα, όσον αφορά τα επιμέρους θέματα, χωρίς να μακρηγορώ, να σταθώ σε δύο σημεία από όλα τα σημαντικά που είπε ο κύριος υπουργό Πρώτα-πρώτα η διαδικασία της ένταξης της ΚΟΣΤΟΝΟΣΑ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει την προσχώρηση της χώρας στον ΟΣΑ. και επίσης η υπηρεσία ευρωπαϊκής εξωτερικής δράσης πρόκειται να συνεργαστεί με τη χώρα. Τώρα βέβαια δεν μπορούμε να συζητήσουμε την οικονομική πτυχή γιατί αυτά είναι άλλα θέματα τις δικές τους λεπτομέρειες αλλά τέλος πάντων θα πρέπει να τονίσουμε το ότι εγκρίθηκε ένα σχέδιο το οποίο χρηματοδοτήθηκε από αυτήν την εταιρική σχέση για διάφορες πολιτικές που είναι σημαντικές για την χώρα. Και πρώτον αναφέραμε την διακυβέρνηση, τη δημόσια, την βιωσιμότητα, επίσης την δημοσιονομική. Και είπαμε ότι για την ένταξη της χώρας των ΟΣΑ πρόκειται για μια μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα, αλλά και για τους εταίρους και φίλους της ε, Κωνσταντίνα. Και έτσι να συνεχιστεί αυτή η φιλόδοξη διαδρομή θεσμικών και νομοθετικών μεταρρυθμίσεων εν κατακλείδη για να θίξω κάτι άλλο σημαντικό για αυτή την ε, Προεδρία της χώρας στη Γραμματεία ΣΥΑΚΑ. Έχουμε πολλές προσδοκίες από αυτή την ε, προσδοκία. Θα έχουμε ευκαιρία όλοι να προχωρήσουμε χέρι-χέρι. Και να υπάρξει μια συνένεση στην Κεντρική Αμερική για μια τέτοια κοινή πορεία. Οπότε και θεωρούμε ότι η περιφερειακή ολοκλήρωση της Κεντρικής Αμερικής είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και για μας και για την περιοχή εκείνη. Εμείς ε, πρεσβεύουμε την περιφερειακή ολοκλήρωση και την υποστηρίζουμε. Αλλά τελικά χώρες Αμερικής θα πρέπει να αποδείξουν την αποφασιστικότητα και βούλησή τους προς τούτο. Οπότε μπορούμε παρά να ευχαριστήσουμε για αυτές τις κοινέ προτεραιότητες της Γραμματείας και της Προεδρίας για τον Παναμά και την Κωνσταντίνα για την πλήρη συμμετοχή σε αυτές τις προσπάθειες όλων των χωρών της Κεντρικής Αμερικής. Και πάλι σας ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ και ευχαριστούμε και εσάς για την ευκαιρία της εκδήλωσης. Και εγώ σας ευχαριστώ κύριε Φόνς και τώρα τον λόγο έχουν οι συνάδελφοι. Ε, τον λόγο έχει ζητήσει ο κύριος Ούρτασουν. Δικό σας. Ε, ευχαριστώ κύριε Υπουργέ που ήρθατε να συναντηθούμε και έχω κάποιες ερωτήσεις για τα όσα μας παρουσιάσατε. Πρώτα-πρώτα σε σχέση με την Προεδρία που ασκείται για την γραμματεία ΣΥΕΚΑ. Η επόμενη χώρα που θα σας δει θα είναι ο Παναμάς και είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί εδώ στο Κοινοβούλιο από την αρχή της θητείας μας για τους μηχανισμούς παγκόσμιας διακυβέρνησης ούτως ώστε να σταματήσει η φοροδιαφυγή, η φοροαποφυγή να δούμε τι θα γίνει και με αυτά τα σκάνδαλα του Panama Gate και έχουμε επίσης και μια ειδική ερευνητική επιτροπή πάνω σε αυτό. Τώρα στα πλαίσια της γραμματείας ΙΕΓΑ είπατε ότι υπάρχει αυτή η διαδικασία του διαλόγου, αυτού του είδους ε, η διεθνής ανταλλαγή πληροφοριών για τα φορολογικά και καλό το ότι ασχολείστε γιατί για εμάς μας απασχολούν αυτά τα ζητήματα Και έχουμε σχετικές συμφωνίες με διάφορες χώρες ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό το οποίο μας καίει ιδιαίτερα όσον αφορά την γεωγραφική περιοχή σας, και αυτό το ξέρετε, είναι το ζήτημα της βίας. Έχουμε ασχοληθεί αρκετά με το θέμα αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να βοηθήσει να υπάρχουν κάποιοι μηχανισμοί αναστολής αυτής της βίας και και είπαμε ότι εσείς είστε μια μικρή οάση μέσα σε μια ζούγκλα βίας. Πέστε μας πάνω σε αυτό. Τι περιφερειακή στρατηγική υπάρχει για το πρόβλημα. Υπάρχει κάποιο άλλο συνάδελφο που θα να θέσει ερώτηση ή όχι. Κύριε Υπουργέ, το λόγο έχετε εσεί. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ε, υποφεληθώ της ευκαιρίας προκειμένου να ευχαριστήσω καταρχήν την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ε, για την βοήθεια που μας έχει παράσχει και την γενεοδορία καθώς επίσης και την αποφασιστικότητά της. να συνδράμει την Κωνσταντίνα στις προσπάθειές της να ενταχθεί στον ΟΣΑ. Ε, πολύ χρήσιμη ε, αυτή η βοήθεια. Σε ό,τι αφορά την ερώτησή σας, κύριε Βουλευτά. Ο ΣΑ ως σημείο αναφοράς και ως ε, οργάνωση που προωθεί ε, μέσω συστημικών μέσων την βελτίωση της παγκόσμιας φορολογικής διακυβέρνησης είναι ε, ένας από τους ε, λόγους ε, που θέλουμε να ενταχθούμε σε αυτόν είναι δηλαδή η ανάγκη τέτοιου είδου συστημικά μέσα φορολογικής διακυβέρνησης να έρθουν και να εφαρμοστούν στην Κεντρική Αμερική. Νομίζω ότι κάθε μία από τις χώρες μας, παρά τις ιδιαιτερότητές τους κάθε μία, θα είχαν να κερδίσουν από την ένταξή τους. Εμείς είμαστε ήδη πολύ προχωρημένοι και ελπίζουμε θα ολοκληρώσουμε τις εργασίες μας φέτος. Έχουμε συζητήσει με, και με τους υπόλοιπους συναδέλφους όμως, για παράδειγμα με τον Παναμά. Οι συνάλφοι του Παναμά ήδη συνεργάζονται με τον ΩΣΑ. Εντατικά θα έλεγα, έτσι ώστε να αναζητηθούν οι μηχανισμοί συμπερίληψης των προδιαγραφών του ΟΣΑ στις δικές του πρακτικές. Το ίδιο θα συμβεί και με τις υπόλοιπες χώρες της Κεντρικής Αμερικής. Συνεπώς αυτό το παράδειγμα διακυβέρνησης. Ε, το παράδειγμα του, του ΟΣΑ θα μπορούσε πράγματι να χρησιμεύσει και ήδη είναι παρόν στις συζητήσεις που λαμβάνουν χώρα. Σε ό,τι αφορά το θέμα της βίας. Δυστυχώς είναι ένα ζήτημα παγκόσμιο. Στην Κεντρική Αμερική το βλέπουμε ήδη ε, Και στην Κολομβία υφίσταται μια διαδικαστική διαδικασία και στο Βόρειο Μεξικό. Ε, αυτές οι διαδικασίες πιέζουν την Κεντρική Αμερική και αυτό που βλέπουμε ήταν προβλεπόμενο. Ε, το θέμα της βίας είναι στην ημερήσια διάταξη των χωρών μας και θα πρέπει η προσέγγιση μας να είναι περιφερειακή. Δεν είναι δυνατόν να είναι κατακαιρματισμένη ένα χώρα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να απασχολήσει όλη την περιοχή μας στην Κεντρική Αμερική και αυτό το θέτουμε στους ε, αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων κατά προτεραιότητα και θα συζητηθεί επανειλημμένων στις ε, ε, διαπραγματεύσεις που θα γίνουν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου μας. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Η κυρία Αντρική αναζήτησε το λόγο και τον έχει αμέσω. Thank you very much, Madam Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαι από την ε, Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Λιθουανή στην καταγωγή. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Για όσα μας εξηγήσατε και Μα ήταν πολύ ενημερωτικά, όλα αυτά μας προβληματίζουν και ποιήσεις από ό,τι ξέρω, βέβαια λόγω της θέσης σας πρέπει να μιλάτε με τρόπο διπλωματικό. Έτσι, πολύ διπλωματικά μας τα είπατε. Αλλά για επεκταθείτε σε παρακαλώ στα εξή. Αυτά που είπε ο συνάδελφος δηλαδή για το TPP. Είδαμε ποιο ήταν το μήνυμα από τη νέα Αμερικανική κυβέρνηση ότι θα πρέπει να ανασταλεί Μεξικό, Χιλή και Περού καλύπτονται. Και εάν λοιπόν ανασταλεί η λειτουργία της συμφωνίας αυτό, πώς θα επιδράσει στην ε, περιοχή σας, τι θα γίνει με την ε, ε, ολοκλήρωση Κεντρικής Αμερικής, ποιος είναι ο μέλλον σχεδιασμός σας τώρα για την ναύτα. Και εδώ είχαμε μια κατηγορηματική δήλωση ότι η ναύτα, η συμφωνία δηλαδή ε, τη Βορειοαμερική είναι το, η χειρότερη εμπορική συμφωνία που γίνει ποτέ. Θα πρέπει να φρενάρει η συμφωνία, θα πρέπει να ανασταλεί η ισχύ τη, θα πρέπει να επαναδιαπραγματευτεί. Και αυτά εσεί πώ τα βλέπετε, πώ θα σα επηρεάσει αυτό όσον αφορά το εμπόριο. Εμεί σε πλευρά Ένωση θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρξει απορρίθμιση και απελευθέρωση του εμπορίου, να γκρεμίσουμε τους στίχους. να άρουμε όλους τους φραγμούς που εμποδίζουν το εμπόριο. Να όμως τώρα που ξεπίδησε αυτή η νέα φιλοσοφία που είναι αντίθετη σε αυτό πιστεύουμε. Ναι, για την ερώτηση κύριε Υπουργέ. Ε, Ευχαριστώ. Για την κυρία Αντρικένεν. Η Λιθουανία και η Κωνσταντίνα είναι δύο χώρες που βρίσκονται στην ίδια διαδικασία ένταξη των ΩΣΑ. Ξεκινήσαμε τις διαδικασίες ένταξη σχεδόν ταυτόχρονα και συναντώμαστε τακτικά με τις λιθουανικές αρχές, ανταλλάσσοντας εμπειρία. Ήταν πολύ σημαντικό που εξελισσόμαστε, είναι σημαντικό που εξελισσόμαστε παράλληλα. Για τις δύο ερωτήσεις που μου θέσατε. Το σε ό,τι αφορά την ε, συμφωνία του ειρηνικού, την TPP. Ε, όπως γνωρίζετε, είναι ένα εμπορικό εργαλείο, μια εμπορική συμφωνία που στόχευε να γίνει το καινούριο πρότυπο, το καινούριο στάνταρ ε, εμπορικών πολυμερών συμφωνιών. στην διαπραγμάτευσή της συμπεριλήφθησαν μια σειρά νέων τομέων και κλάδων ε, και ο, το εμπόριο του 21ου αιώνα ε, δεν χαρακτηρίζεται από ψηλούς δασμούς. Οι περισσότερες χώρες έχουν χαμηλούς δασμούς. Το θέμα λοιπόν δεν είναι εκεί στην κατάργηση των δασμών. Είναι στην διευκόλυνση του εμπορίου, στην κατάργηση των φραγμών και των εμποδίων. Στην κατάργηση των εργαλείων πολλές φορές χρησιμοποιούνται για να μπλοκαριστεί το εμπόριο. Συνεπώς, το πλεονέκτημα που βλέπαμε εμείς σε αυτή τη συμφωνία ήταν ότι είχε το θάρρος να πάει λίγο πιο μακριά και να προτείνει καινούριε προδιαγραφέ, Μια καινούρια δηλαδή γενιά συμφωνιών να δημιουργήσει. Εμεί δεν ήμασταν βέβαια τμήμα των αρχικών διαπραγματεύσεων και καμία χώρα τη Κεντρική Αμερική δεν συμπεριελήφθη, αλλά παρακολουθούσαμε πολύ στενά και με πολύ ενδιαφέρον τι διαπραγματεύσει αυτέ. Την TPP δεν την πρότειναν μεγάλε χώρε, αλλά μικρέ. Το Μπρουνέι, η Νέα Ζηλανδία κλπ. Είναι χώρε πιο μικρέ Οπότε είναι σημαντικό να το δούμε από τη δική του πλευρά. Βέβαια, η TPP ε, θα πληγεί αν οι Ηνωμένε Πολιτείε αποχωρήσουν, διότι θα διακοπεί αυτή η διαδικασία συζήτησης και διαπραγμάτευσης που ε, είχε ως στόχο να ξεπεράσουμε τα παραδοσιακά και να δημιουργήσουμε μια καινούργια γενιά συμφωνιών που θα ξεπερνάει την απλή κατάργηση των δασμών. Δεν ξέρουμε τι θα συμβεί βέβαια. Στην τελευταία σύνολο κορυφής ΑΠΕΚ, ο, ο πρόεδρος της Κίνας είχε πει ότι ενδεχομένως η Κίνα θα ενδιαφερόταν να ενταχθεί. Στην άτυπη συνεδρία Υπουργών Εμπορίου στον Ταβό πριν από δύο εβδομάδε, οι συνάδελφοι από την, τον Καναδά, την Ιαπωνία, την Νέα Ζηλανδία και την Αυστραλία άνοιξαν τα αυτιά τους και άρχισαν να σκέφτονται την δυνατότητα η TPP να αναπτυχθεί ως συμμαχία του ειρηνικού με καινούρια μέλη. Ε, η διαδικασία συμμαχίας του ειρηνικού έχει τεράστια σημασία η Χιλή, το Περού, η Κολομβία και το Μεξικό συμμετέχουν. Η Κοσταρικά είναι αυτή τη στιγμή υποψήφια χώρα ένταξης στη Συμμαχία του Ειρηνικού. Ε, εξετάζουμε διάφορα σενάρια, διάφορες δυνατότητες διαπραγμάτευσης με την Συμμαχία για τον Ειρηνικό και ε, σε αυτό το πλαίσιο έχουμε εντοπίσει μια σειρά δυνατοτήτων. Η Συμμαχία για τον Ειρηνικό δεν είναι μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου. Είναι μια διαδικασία ολοκλήρωσης. Φιλόδοξη διαδικασία ολοκλήρωσης και το ενδεχόμενο ένταξης δεν αφορά μια συμφωνία ε, ελεύθερου εμπορίου αλλά μια συμφωνία, μια πρωτοβουλία ε, ένταξης. Θα πρέπει να αναλύσουμε βέβαια το πώς θα γίνει μια τέτοια ένταξη. Είναι αυτά η Συμφωνία Ελεύθερων Εμπορίου Βορεια Αμερική. Εδώ είναι σημαντικό να διευκρινίσουμε το εξή. Το Μεξικό, οι Ηνωμένε Πολιτείε και ο Καναδά ε, έχουν εμπορικές σχέσεις στο πλαίσιο τη ναύτα. Είναι μια συμφωνία του 1993, πριν τη δημιουργία του ΠΟΕ δηλαδή, του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Είναι λοιπόν μια συμφωνία παλιά γενιά. Μια αναδιαπραγμάτευση αυτή της συμφωνίας θα μπορούσε ενδεχομένω να οδηγήσει στην ένταξη καινούριων τομέων ή καινούριων μέσων και ενδεχομένως θα ήταν καλό για τα τρία μέρη. Δεν ξέρω αν αυτή είναι η, πρόθεση, έτσι, δεν είναι σαφές. Μέχρι να το διευκρινίσουμε δεν είναι δυνατόν να λάβουμε θέση. Τώρα, η Κεντρική Αμερική μαζί με την Δομινικανή Δημοκρατία είναι χώρες της ΣΥΕΚΑ. Έχουμε δηλαδή εμείς στη διάθεσή μας άλλο ε, όργανο που είναι η ΚΑΦΤΑ, η ε, Συμφωνία Ελεύθερων, Ελεύθερων Πορείου Κεντρικής Αμερικής. Από το 2007. Είναι πιο νέα συμφωνία. Τελευταίας δεκαετίας. Η κάφτα σε σχέση με την ναύτα έχει την εξή διαφορά. Η ναύτα ε, για τις ε, Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια συμφωνία που οδηγεί σε εμπορικό έλλειμμα. Και αυτό το εμπορικό έλλειμμα είναι που πυροδοτεί τις δυσκολίες. Στην περίπτωση της κάφτα. Η κάφτα είναι μια συμφωνία ε, πλεονασματική για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν λοιπόν το πρόβλημα των ΗΠΑ είναι τα πλεονάσματα, τα ελλείμματα, η καύτα δεν τους δημιουργεί έλλειμμα, άρα ενδεχομένως δεν του δημιουργεί και προβλήματα. Η ναύτα από την άλλη μεριά ε, στηρίζεται πολύ στην βαριά βιομηχανία. Αυτός είναι ένας κλάδος στον οποίο οι ΗΠΑ έχουν σημαντικά προβλήματα παραγωγικότητας γιατί σε ένα μεγάλο βαθμό βαριά βιομηχανία έχει μετακινηθεί εκτός των ΗΠΑ. Στην περίπτωση της ΚΑΦΤΑ, μεταξύ Κεντρικής Αμερικής και ΗΠΑ, ε, το εμπόριο εστιάζεται κυρίως στο γεωργικό τομέα, στον αγροτικό τομέα. Κυρίως αγροτικά προϊόντα τα οποία δεν παράγουν οι ΗΠΑ. Οπότε εκεί υπάρχει μια θεμελιώδης διαφορά μεταξύ της ΝΑΦΤΑ και της κάφτα καταλαβαίνουμε γιατί η ναύτα δημιουργεί τα συγκεκριμένα προβλήματα και γιατί η καύτα ενδεχομένως δεν θα ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο. Το πώς θα επηρεαστεί το εμπόριο μεταξύ, μάλλον το πώς επηρεάζουν οι ΗΠΑ το εμπόριο της Ρίκα. Η Κώστα Ρίκα είναι από τις χώρες που έχουν τη μικρότερη εξάρτηση από τις ΗΠΑ. Το 36% των εξαγωγών μα πηγαίνουν στι ΗΠΑ, αλλά υπάρχουν άλλε χώρε τη Κεντρική Αμερική που περισσότερο το 50% των εξαγωγών του προορίζονται για τι ΗΠΑ. Ε, τώρα, οι επενδύσει όμω είναι ψηλέ. Οι επενδύσει των ΗΠΑ είναι ψηλέ στην Κεντρική Αμερική. Σε εμά βέβαια είναι κάτω από το 40%. Σε άλλε χώρε είναι ακόμα μεγαλύτερο. Οπότε εμεί εξαρτώμεθα λιγότερο από τι ΗΠΑ. Απ' την άλλη μεριά έχουμε και τα εμβάσματα τα εμβάσματα των πολιτών μας που ζουν στο εξωτερικό. Σε ορισμένες χώρες της Κεντρικής Αμερικής αυτά τα εμβάσματα αντιπροσωπεύουν το πάνω από το 15% του ΑΕΠ. Οπότε ε, τέτοιου τύπου δράσεις σε σχέση με το μεταναστευτικό μπορεί να επηρεάσουν πολύ αυτές τις χώρες. Σε εμά ε, τα εμβάσματα είναι πολύ μικρότερα. Αντιπροσωπεύουν ένα πολύ μικρότερο ποσοστό του ΑΕΠ μας. Όμως το πρόβλημα είναι περιφερειακό. Ορισμένες περιοχές μπορεί να, ορισμένες χώρες μπορεί να επηρεαστούν περισσότερο και άλλες λιγότερο, αλλά γενικά η περιοχή μας θα επηρεαστεί. Εγώ ζητώ από τους, ζήτησα από τους υπουργούς ε, οικονομίας της Κεντρικής Αμερικής να, να συναντηθούν για να συζητήσουν αυτό ακριβώς το θέμα και τις συνέπειες των αποφάσεων των ΗΠΑ. Πρέπει να τις παρακολουθήσουμε με πολύ προσοχή. Κύριε συνάδελφοι, υπάρχει άλλη ερώτηση. Όχι. Κυρία Κινίτση, αντιπρόεδρος της Επιτροπής μας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, να σας τα πω στα Ιταλικά μια που έχουμε τους διερμηνείς. Ευχαριστώ του συμπροέδρους, ευχαριστούμε και τον κύριο Υπουργό για τα όσα μας παρουσίασε. Ε, βέβαια, και συμφωνώ με την υπόθεση της ένταξης της ε, χώρας στον ΟΣΑ. Τα είπαμε σχετικά με αυτό το σημείο, αλλά εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Τι γίνεται με αυτό το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, ποιους τομείς θα καλύψει, τι προσδοκάτε από αυτές τις αλλαγές και μιλώ για νομοθετικές μεταρρυθμίσεις πολιτικές κοινωνικές προνοίας, πολιτικές ε, υγείας και τον εργασιακό τομέα. Καλά, έχουμε και το θέμα της βίας πολλών μορφών, αλλά τι θα γίνει επίσης και με το θέμα της παιδείας, γιατί υπάρχουν κάποιοι ανήλικοι, ιδίω κάποια βρέφη που ξέρουμε ότι βρίσκονται σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, χρειάζονται υποστήριξη μέσω κάποιων κοινωνικών πολιτικών. Αυτό πρέπει να το προσέξετε. Οπότε, αν μπορείτε, πέστε μας δύο λόγια πάνω σε αυτό. Τι γίνεται με τα ρυθμίσει που έχετε αρχίσει. Και επίσης, τι αποτελέσματα προσδοκάτε να αποσπάσετε από αυτές τις αλλαγές. Κύριε Υπουργέ, θα σας δώσω το λόγο να απαντήσετε. Θα σας παρακαλούσα όμως σύντομα, γιατί ο χρόνος μας τελειώνει. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό για τους διερμηνείς μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε για την ε, ευκαιρία μου δίνετε να θίξω αυτό το θέμα. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις που έχουμε αρχίσει επειδή τη του ΩΣΑ αφορούν πολλούς τομείς. Έχουμε εδώ δύο βασικούς άξονες. Πρώτα-πρώτα η νομοθετική μεταρρύθμιση και η διοικητική. Η πρώτη αφορά το κοινοβούλιο, η δεύτερη την κυβέρνηση. Και αυτή η δυναμική του ΩΣΑ έχει ως εξής Έχουμε διάφορες επιτροπές που έχουν κάνει κάποιες ε, μελέτες για διακρύβωση της κατάστασης στη χώρα και κάθε επιτροπή ορίζει κάποιες μεταρρυθμίσεις. Σήμερα έχουμε 20 μελέτες οι οποίες ολοκληρώνονται ε, ολοκληρώθηκε σχετική μελέτη για το εμπόριο άρα επομένως ε, έχει ενεργοποιηθεί αυτή η διαδικασία. Τώρα το θέμα της ε, δημόσιας υγείας, πολύ σημαντικό, η βιωσιμότητα του συστήματος που έχει η χώρα όσον αφορά τη δημοσία υγεία. Όλοι καλύπτονται στη χώρα. Αλλά είναι τώρα θέμα ποιότητας και βιωσιμότητας. Αυτό μας απασχολεί και για τις συντάξεις έχουμε ένα σύστημα για να καλύπτονται όλοι και εδώ μας απασχολεί η βιωσιμότητα αυτών. Όσον αφορά την ε, παιδεία, θα πρέπει να μελετήσουμε το θέμα της ε, ποιότητα. Πρόσφατα ξεκίνησε με κάποια στεγνωτική μεταρρύθμιση το ότι έχει υποχρέωση το κράτος να επενδύει τουλάχιστον το 8% του ΑΕΠ για την ε, ε, δημόσια παιδεία. Πολλά λεφτά. Αλλά ακριβώ, προς τα εκεί, σε συνεργασία με τον κινούμεθα. Τώρα για την κοινωνική πολιτική έχουμε τώρα μπει στο να κάνουμε κάποια καταγραφή του πληθυσμού. Πάμε έχουμε δύο τρίτα γυναίκες, οπότε οι γυναίκες που εντάσσουν στην αγορά εργασίας είναι δύο στους τρεις που τα τελευταία 20 χρόνια έχουν μπει στην αγορά εργασίας. Άρα θα πρέπει να βρούμε ένα πρόγραμμα να καλύψουμε τους πιο ηλικιωμένους αλλά και τους ανήλικους γιατί έτσι θα βοηθήσουμε τις γυναίκες να ε, αναπτύξουν επαγγελματική δραστηριότητα. Ε, επίσης είπαμε ότι θα κάνουμε και κάποιες ε, φορολογικές ε, μεταρρυθμίσεις σε συνεργασία με τον ΩΣΑ. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ και τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Πρόεδρο, στον κύριο Μπόγκε, να συνοψίσει τα τελικά συμπεράσματα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μωρά, για αυτή την ανταλλαγή απόψεων. Πολύ ενδιαφέρον τόσο μας εξηγήσατε. Όσον αφορά το ελεύθερο εμπόριο, πολλές φορές στην Ευρώπη θεωρούμε ότι ελεύθερο εμπόριο σημαίνει αχαλήνωτη απορρίθμιση χωρίς κανόνες, χωρίς πρότυπα. Όμως σωστά είπατε ότι οι σημερινές εμπορικές συμφωνίες δεν αφορούν τόσο πολύ των δασμών, αλλά τα άλλα, τα μη δεσμολογικά θέματα, ήδη στο παρελθόν έχουν γίνει πολλά για τους δασμούς. Όμως, θα πρέπει να κερδίσει κανείς την πλειοψηφία του κόσμου και για το πετύχει αυτό θα πρέπει κάποιος να εξηγήσει ότι δεν πρόκειται ε, για το ότι αυτό σκοπός είναι το ελεύθερο εμπόριο αλλά κοινέ αξίες και το ότι προσπαθούμε να έχουμε μια νέα γενιά εμπορικών συμφωνιών επί τη βάση συγκεκριμένων κανόνων. Όντως πολλές φορές γίνονται προσαρμογές και διορθώσεις, αλλά είναι πολύ σημαντικό να κερδίσει κανείς την κοινή γνώμη όσον αφορά την παγκοσμιοποίηση. Επίσης, σε εύχομαι καλή επιτυχία σε αυτό το πρόγραμμα δράσης όσον αφορά την Τελωνιακή Ένωση. Θα παρακολουθήσουμε με ενδιαφέρον τις προσπάθειές σας γιατί είναι σημαντικό βήμα πρόοδου για αυτή την περιφερειακή συνεργασία και την οικονομική ολοκλήρωση. Και αυτό αφορά και την προσπάθειά σας μέχρι το 2018 να έχετε γίνει μέλος του ΟΣΑΚΑΤΗ το οποίο νομίζω θα είναι θετικό, θα είναι παράδειγμα προσμήμιση και για άλλες χώρες. Τέταρτο που θέλω να σας αναφέρω, ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα οποία μας είπατε όσον αφορά αυτήν την ψηφιακή εμπορική πλατφόρμα. Πριν από μια πενταετία ήμουν στην Αργεντινή και πέρσι στην Χιλή και κατάλαβα ότι η ελεύθερη πρόσβαση στο ίντερνετ ε, σε κάποιες ε, μεσαίου μεγέθους πόλη σε κάποια ξενοδοχεία της σειράς ήταν πιο αποτελεσματική από ό,τι στη δική μου χώρα. Άρα αυτού του είδους η ψηφιοποίηση είναι βασική πρόκληση όπως παντού στον κόσμο. Αλλάζουν οι μεθοδολογίες, αλλάζουν όλα. Και ε, από οικονομικής πλευράς, από κοινωνικής πλευράς. Αυτές οι πλατφόρμες, οι ψηφιακές. Το, το ότι κάποιος θα πρέπει να χρησιμοποιεί την καλύτερη από τις υπάρχουσες τεχνολογίες. Να ποιε θα είναι οι εξελίξεις οι οικονομικές στο μέλλον. Και πάλι ευχαριστούμε για την ευκαιρία να συζητήσουμε σήμερα και καλή επιτυχία στην ε, Προεδρία που έχετε. Uh, uh, λοιπόν, κλείνοντας, να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου τον κύριο Υπουργό για την ε, εξαιρετική τοποθέτηση που είχε και τις πληροφορίες που μας έδωσε, την υπέροχη συζήτηση που ακολούθησε και το ενδιαφέρον των συναντέλφων με τις ε, ε σημαντικές ερωτήσεις που κάνανε, να ευχαριστήσω όλα τα μέλη των διπλωματικών αποστολών, τα μέλη των ε, θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους συναδέλφους που ήταν σήμερα εδώ σε αυτή τη συζήτηση και είναι πολύ σημαντικό αυτό για μας ε, όπως επίσης θα μου επιτρέψετε να τελευταίως να κλείσω με, τα, με τους ε, κυρίους κυρίους μεταφραστές οι οποίοι πάντα δείχνουν μια ανοχή στι επιτροπές μας και μας ε, συμπαραστέκονται όταν καθυστερούμε τόσο πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.